Ετοιμάζουμε την ε, συνεδρίαση του Συμβουλίου ε, στις 21 και 22 ε, Μαρτίου για τον Brexit. Η κυρία Σότ, εκ μέρους του Συμβουλίου, έχει το λόγο. Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε διαπραγματευτεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχει μια σειρά συζητήσεων ε, για μια σειρά προκλήσεων ε, που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας ξεκινήσω από την, Ευρωπαϊκή, από την οικονομία. Οι ε, ευρωπαϊκοί ηγέτες θα συζητήσουν την οικονομία και το 19ο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Η Ευρώπη, όπως και ο υπόλοιπος κόσμος, αντιμετωπίζει συστημικές αλλαγές ε, όπως είναι η ψηφιακή ε, μετάβαση, η οικονομία των δεδομένων και η μετάβαση σε μια πιο πράσινη οικονομία. Το να ελέγξουμε αυτέ τι ευκαιρίε, το να αδράξουμε αυτέ τι ευκαιρίε, θα είναι το κλειδί για την μελλοντική μα ευημερία. Για να ενισχύσουμε την οικονομική μα βάση θα πρέπει να φροντίσουμε οι πολιτικέ μα. η ψηφιακή, η βιομηχανική, η εμπορική είναι εναρμονισμένε ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτέ τι προκλήσει και να προωθήσουμε τα στρατηγικά συμφέροντα τη Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα έχει μια οριζόντια συζήτηση για το θέμα αυτό. Άλλο κρίσιμο θέμα είναι η αλλαγή του κλίματος, το οποίο μόλις συζητήσαμε. Όπως ε, σημειώθηκε στη συζήτηση αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να γίνει πιο φιλόδοξη και να συνεχίσει να ηγείται στην κλιματική δράση. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί το ισχύον πλαίσιο 2030, αλλά να ε, επενδύσει και σε μια μακροπρόθεσμη μετάβαση σε ε, μια οικονομία φιλική προς το κλίμα. Θα πρέπει να φροντίσουμε να μην μείνει κανείς πίσω. Ε, να, λαμβάνοντας υπόψη περιφερειακές ιδιαιτερότητες και διάφορες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συζητήσει το θέμα αυτό και θα, ε, ε, και θα δημιουργήσει τον προσανατολισμό για τα θέματα αυτά. Η Κίνα είναι πολύ σημαντικός παράγοντας και οι ηγέτες θα συζητήσουν τις σχέσεις μας με την Κίνα και τέλος, ε, θεμελιώδης λίθος ε, της οικονομίας μας είναι οι πολίτες να μπορούν ε, να ψηφίζουν με τρόπο ασφαλή και με βάση τα γεγονότα. Θα αναφερθούν λοιπόν οι τελευταίες εξελίξεις για προστασία της δημοκρατικής διαδικασίας από χειραγώγηση εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ηγέτες θα ενημερωθούν σχετικά με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες ε, στον τομέα αυτών, ακολουθώντας το ε, κοινό σχέδιο δράσης που παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ύπατη ε, εκπρόσωπο τον Δεκέμβριο. Επίσης ε, θα συνεδριάσει υπό τη σύνθεση του άρθρου 50 ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να συζητήσει το Brexit. Πρόεδρε, ε, κύριοι και κυρίες ευρωβουλευτές, να ζει κανείς ή να μην ζει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υπάρχει ή να μην υπάρχει. Αυτό θα πρέπει να συζητήσει το Βρετανικό κοινοβούλιο και δεν βρισκόμαστε εδώ στη σκηνή, στο θέατρο. Μιλάμε για την πραγματική ζωή και σε αυτήν την ύστερη φάση καλούμεθα να διευκολύνουμε την ε, εφαρμογή της συνθήκης αποχώρησης που συμφωνήθηκε πέρσι, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να είναι εις βάρος της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, ιδιαίτερα όσον αφορά την Ιρλανδία με τις πρόσθετες διασφαλίσεις που δώσαμε τον ε, Δεκέμβριο, το Ιανουάριο και την Δευτέρα είναι πολύ δύσκολο να δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Όχι μόνο όσον αφορά τα δικαιώματα των πολιτών ε, και, ε, και τον Ιρλανδικό Μηχανισμό Ασφαλείας, το backstop, πρέπει να μην αμφισβητήσουμε την ε, ανάγκη του backstop. Ε, υπάρχει όμως η επιθυμία να είναι προσωρινό μέτρο. Από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουμε να προωθήσουμε τα συμπεράσματα και πιστεύουμε ότι μέσα σε λίγες μέρες θα έχουμε κάποια λύση εφόσον η Βρετανική πλευρά ξεκαθαρίσει τι θέλει. Είναι όμως πάρα πολύ πιθανό, ακόμα και αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψηφίσει την ε, συμφωνία αποχώρησης μέσα στις επόμενες μέρες, ε, η απόφαση αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από έκκληση για παράταση χρονική. Αυτό σημαίνει προσαρμογή της ε, συμφωνίας ε, και καθυστέρηση της διαδικασίας, η οποία θα πρέπει να συμφωνηθεί από το επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Κατά την εξέταση ενός τέτοιου αιτήματο ε, θα ζητήσουμε ε, αξιόπιστη ε, αιτιολόγηση για την διάρκεια και τον στόχο μιας παράτασης. Πιστεύω όμως ότι τα θεσμικά όργανα θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν με καλό τρόπο την διαδικασία αυτή, ώστε να έχουμε μια έγκαιρη εφαρμογή της συμφωνίας. Όπως σας είπα και πριν, είμαστε ανοιχτοί για συζήτηση εφόσον ε, δεν χάνουμε από τα μάτια μας τον στόχο των συζητήσεων αυτών. Το... Η κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να δείξουν την κατεύθυνση προς την οποία θέλουν να προχωρήσουν και μάλιστα με σχετικό χρονοδιάγραμμα. Στο μεταξύ, η μόνη βεβαιότητά μας είναι η αυξανόμενη αβεβαιότητα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ε, και με σαφή οικονομικό αντίκτυπο στις επενδύσεις και ακόμη πιο σημαντικά στις θέσεις απασχόλησης. Γι' αυτό είναι όλο και πιο απαραίτητο να προετοιμαζόμαστε για κάθε ενδεχόμενο ε, συμπεριλαμβανομένη της αποχώρησης χωρίς συμφωνία. Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη σε εθνικό επίπεδο ε, προετοιμάζονται και βασίζονται στην δουλειά που ήδη έχει γίνει τώρα. Τα μέτρα ετοιμότητας ε, και προετοιμασίας ε, των ε, θεσμικών οργάνων με κάνουν αισιόδοξη. Η Προεδρία είναι πεπισμένη ότι με τη δική σας συνεργασία θα μπορέσει να ολοκληρώσει την υιοθέτηση των ε, μέτρων που απομένουν. Ταυτόχρονα ελπίζουμε ότι δεν θα είναι απαραίτητα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Τσότ. Τώρα ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Τίμερμανς. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να είμαστε λοιπόν μετά από ακόμα μία ψηφοφορία στη Βουλή των Κοινοτήτων. Έχει καταψηφιστεί η Συμφωνία Αποχώρησης. Ε, παρά τις επιπρόσθετες διευκρινήσεις που δόθηκαν, παρά των τεράστιων προσπάθειων που κατέβαλαν ε, ο κύριος Μπαρνιέ και ο κύριος Γιούνκερ για να βοηθήσουν την κυρία Μέη να διευκρινίσει τα ζητήματα που εκκρεμούν και πάλι όμως καταψηφίστηκε η συμφωνία. Και πάλι λοιπόν σήμερα θα περιμένουμε την επόμενη ψηφοφορία στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Γιατί ο μόνος που μπορεί να μας δώσει κάποια κατεύθυνση για το πού θα πάμε από εδώ και πέρα είναι οι Βρετανοί βουλευτές. Και πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθούν την ίδια προσέγγιση. Να βλάψουν όσο γίνεται λιγότερο του Ευρωπαίου. Είτε μένουν στο Ηνωμένο είτε στην Υπηρετική Ευρώπη. Αυτό είναι το δικό μα καθήκον και μέλημα. Να σκεφτούμε του πολίτε μα, ε, τι επιχειρήσει μα, τα συμφέροντά μα και από τι δύο πλευρέ ε, τη μάχη. Και το λέω αυτό γιατί αυτό που κατά βάση προσπάθησα να κάνω και εγώ αλλά και ο Μισελ είναι να διασφαλίσουμε ότι οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει η Βρετανική κυβέρνηση και η δική μας ανάγκη να αποφύγουμε ένα πραγματικό σύνορο στην Ιρλανδία και να διασφαλίσουμε την ακαιρεότητα της εσωτερικής αγοράς, κάπως θα συγκεραστούν. Εγώ δεν βλέπω κάποια καλύτερη λύση από τη συμφωνία αποχώρησης μαζί με όλες τις διευκρινήσεις που δόθηκαν. Αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση σήμερα. Φυσικά και θα συνεχίσουμε ε, αυτή την προσέγγιση να κάνουμε όσο γίνεται λιγότερη ζημιά σε μια πολύ επιζήμια διαδικασία. Γιατί το Brexit είναι κάτι το ιδιαίτερα επιζήμιο και για το Ηνωμένο Βασίλειο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά είναι δικό μα καθήκον, βάσει τη ε, ψήφου των ε, Βρετανών πολιτών, να προχωρήσουμε σε ένα Brexit όσο γίνεται λιγότερο επιζήμιο. Δεν θα αλλάξει λοιπόν αυτό. Σήμερα όμω βρισκόμαστε στα χέρια του Βρετανικού πολιτικού συστήματο. Εκείνοι πρέπει να μα πούν τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Η λύση θα έρθει από το Λονδίνο και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Υπάρχουν και άλλα θέματα που πρέπει να διαχειριστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επικεντρώνεται και σε άλλα ζητήματα. Βιομηχανική πολιτική. Η βιομηχανία μας είναι ισχυρή και είναι ε, κινητήριο μοχλός ε, της οικονομίας μας. Δίνει δουλειά σε 32 εκατομμύρια πολίτες ε, και αποτελεί τα δύο τρίτα των εξαγωγών μας. Έχουμε πολλούς εταίρους που μας χτυπούν την πόρτα για να διασφαλίσουν ελεύθερες συναλλαγές. Όμως πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Πρέπει να ενισχυθούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με το δίκαιο ανταγωνισμό εντός της Ένωσης και με μια ηγετική θέση σε διακυβεύματα όπως η κλιματική αλλαγή. Έχουμε μείζονο σημασία πολιτικά προγράμματα, ε, συσσωρευτέ ε, νέα γενιά για την ε, καθαρή ενέργεια ή τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα. Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι καθώ ε, εξελίσσονται οι τεχνολογίε, εμεί θα συνεχίσουμε να προασπίζουμε τι αξίε μα. Γιατί τελικά όλα αυτά τα το κάνουμε για να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών. Γι' αυτό θέλουμε ε, αξιοπρεπεί εργασία με ισότιμη μεταχείριση, και ούτω καθεξής. Γι' αυτό καταβάλουμε συστηματικές προσπάθειες να εμβαθύνουμε ε, και να καταστήσουμε πιο δίκαιη την εσωτερική αγορά. Και να αξιοποιήσουμε περαιτέρω τις δυνατότητες που έχουμε στις υπηρεσίες, στην ψηφιακή αγορά και το πολύ σημαντικό στις, ε, στις κεφαλαγορές. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία να εξετάσουμε τι σχέσει μα με την Κίνα, εν ώψη και τη ε, Συνόδου Κορυφή με την Κίνα. Είναι ε, ένα στρατηγικό εταίρο ε, και άλλο έτερο μέλο διαπραγματεύσεων. Προωθεί διαφορετικά μοντέλα διακυβέρνηση. Οι κινέζικε αρχέ έχουν εκφράσει την βούλησή τους ε, να ακολουθήσουν ένα άλλο μοντέλο πιο ανοιχτό και πιο συμπεριληπτικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία από τις πιο ε, ανοιχτές οικονομίες ε, στον κόσμο, αλλά παράλληλα υπερασπίζεται την πολυμέρεια βάσει αξιών που θα είναι ίδια για όλους και θα ακολουθούνται από όλους δεν θα πρέπει να έχουμε μια ε, αφελή προσέγγιση των ελευθέρων συναλλαγών. Γι' αυτό και προτείναμε τη θέσπιση ενό διεθνούς μηχανισμού ε, για τις, ε, για τις δημόσιες προμήθειες σε όλο τον κόσμο. Είναι λοιπόν μια αμοιβαία προσπάθεια, ούτω ώστε να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και συνεργασία με την Κίνα, μεγαλύτερη αμοιβαιότητα, ούτω ώστε και οι επενδυτέ και οι επιχειρήσει μα να επωφελούνται και στην Κίνα των ίδιων συνθήκων και όρων ανοίγματο τη αγορά που προσφέρεται αυτή τη στιγμή στου Κινέζου επενδυτέ στην Ευρώπη. Που δυστυχώ αυτό δεν γίνεται. Έχουμε λοιπόν την υποχρέωση να υπερασπίσουμε τα ε, συμφέροντά μα, ε, τη βιομηχανία μα, του εργαζόμενου και του πολίτε μα ε, από κάθε προσπάθεια του ανταγωνισμού. Πρέπει να φιλτράρουμε τι ε, ξένε επενδύσει για να προστατεύσουμε τα στρατηγικά συμφέροντα τη ε, Ένωση. Χαιρετίζω ε, τις ε, προσπάθειες ε, του Ευρωκοινοβουλίου για μια υιοθέτηση των προτάσεων σε χρόνο ρεκόρ. Θέλουμε να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε το σημερινό, το ισχύον σύστημα πολυμέρειας σε ό,τι φορά και τις κρατικές επιχορηγήσεις. Πρέπει και η Κίνα να αναλάβει το δικό της μερίδιο ευθύνης. Η πραγματική και όσον αφορά την πραγματική κυριαρχία, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει ε, να είναι πρωτοπόρος ε, στο θέμα αυτό. Και η ευθύνη για τους κλιματικούς στόχους σημαίνει για την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο να ε, λαμβάνει υπόψη τους στόχους αυτούς και να επενδύσουμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης, να μην αφαιρέσουμε από κανέναν το εισόδημά του, το οποίο σημαίνει να ε, ενθαρρύνουμε την καινοτομία και να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης υψηλής ποιότητας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις προτάσεις σας, ε, για τις οποίες νομίζω ότι μπορείτε να είστε περήφανοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει ηγετική θέση και να Έχουμε ιδιωτικές επενδύσεις που να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Παρισιού. Με συγκινεί το ότι πολλοί νέοι διαδηλώνουν στους δρόμους για πιο φιλόδοξους στόχους. Μια τέτοια Ευρώπη μου δημιουργεί αισιοδοξία για το μέλλον. Ευχαριστώ την Κρέτα και όλους τους άλλους νέους για την έμπνευση που μας δίνουν. Χρειαζόμαστε τόλμη για να αντιμετωπίσουμε και μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη δημοκρατία μας, τις ηθελημένες ε, προσπάθειες χειραγώγησης του διαλόγου. Το μήνυμά μας είναι ότι η Ευρώπη παραμένει ανοιχτή. Ε, ελευθερία λόγου είναι ε, ένα από τα σημαντικότερα αγαθά μας. Γνωρίζουμε όμως ότι υπάρχουν δυνάμεις που θέλουν να υπονομεύσουν ε, τη δημοκρατία μας και αυτό στον προεκλογικό αγώνα θα είναι μεγάλη πρόκληση. Θα πρέπει λοιπόν να το προσέξουμε. Επικροτώ το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη στηρίζουν τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της παραπληροφόρησης. Βρισκόμαστε όμως μόλις στην αρχή, απομένουν πολλά να γίνουν στον τομέα αυτόν. Κυρίαρχη θα παραμείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο εάν είναι ασυμβίβαστη όσον αφορά τις αξίες μας εντός και εκτός της Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Πρώτη Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τώρα θα δώσω το λόγο στον διαπραγματευτή μας Μισελ Μπαρνιέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους σας. Ιδιάζουσα μέρα σήμερα, σοβαρές υποθέσεις είναι να εξελίξει. στο τέλος αυτής της ε, μακράς διαδικασίας των διαπραγματεύσεων. Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας πω ότι εξ ονόματος της ομάδας ε, που, της οποίας ηγούμε χάρη στην εμπιστοσύνη του Προέδρου Γιούνκερ, ότι είμαι ευγνώμων. Αισθάνομαι ευγνωμοσύνη για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει το Κοινοβούλιο και το είπα προηγουμένως και στη διάσκεψη των Προέδρων ότι αυτή η εμπιστοσύνη δεν πέφτει εξ ουρανού, δεν είναι τεχνητή, δεν δίδεται ως επιταγή εν λευκό. Είναι μια εμπιστοσύνη που βασίζεται στο διάλογο, στη διαφάνεια από την πρώτη μέρα. και η εμπιστοσύνη θα παραμείνει στηρισμένη, θα στηρίζεται πάντα στην ε, εμπιστοσύνη και στο διάλογο. Και η υπουργό και ο κύριος Τίμερμαντς είπε ότι βαραίνει πάνω μας μια φοβερή αβεβαιότητα που δημιουργήθηκε πριν από τρία χρόνια από την κυρίαρχη απόφαση την οποία σεβόμαστε παρότι λυπούμεθα την απόφαση λοιπόν του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η αβεβαιότητα πλήττει και, την, και το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βόρεια Ιρλανδία ιδίω, αλλά κάθε μία από τις ευρωπαϊκές χώρες και εμάς τους ίδιους. Η ευθύνη της απόφασης του Brexit ανήκει αποκλειστικά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και σήμερα η πρώτη ευθύνη για να βγούμε από το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται αυτή η διαπραγμάτευση, η πρώτη ευθύνη ανήκει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το υπενθύμησε πολύ έντονα χθε το βράδυ, αμέσως μετά την ψηφοφορία, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλτ Τούσκ. Προσπαθήσαμε μαζί να βρούμε λύσεις για κάθε πρόβλημα. Και είναι άπειρα τα προβλήματα ανθρώπινα, κοινωνικά, τεχνικά και νομικά, οικονομικά και χρηματοπιστωτικά που δημιουργούνται από τον Brexit. Για να διαχειριστούμε όλες τις συνέπειες, ούτω ώστε να συνοδεύσουμε, γιατί αυτή είναι η γραμμή μας από την αρχή και θα παραμείνει η δική μας αρχή, να συνοδεύσουμε και να πλαισιώσουμε το Ηνωμένο Βασίλειο σε μια έφτακτη αποχώρηση. Από την πρώτη στιγμή της διαπραγμάτευσης, ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να μειώσει αυτή την αβεβαιότητα, εξασφαλίζοντας μία έφτακτη αποχώρηση και χάρη σε αυτή την έφτακτη αποχώρηση και στην βάση εμπιστοσύνη που δημιουργούμε χάρη σε αυτή την έφτακτη αποχώρηση να χρησιμοποιήσουμε τον απαραίτητο χρόνο που θα είναι από 21 μήνες μέχρι 4 χρόνια, όχι παραπάνω, για μια άλλη διαπραγμάτευση. Γιατί πάντα είχα πει ότι είναι η πιο σημαντική, πέρα από τον Brexit είναι ο διαχωρισμός και η μελλοντική σχέση που θέλουμε να χτίσουμε με το Ηνωμένο Βασίλειο, που θα παραμείνει προφανώς μια χώρα φιλική, σύμμαχη και μια χώρα εταίρος. Αυτά κάναμε διαπραγματευόμενοι επί με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και ποτέ εναντίον της Βρετανικής κυβέρνησης. Μια συμφωνία αποχώρησης η οποία θα είναι προς το συμφέρον των πολιτών, των επιχειρήσεων και όλων των ενδιαφερομένων και συμμετεχόνων από τη μία και την άλλη πλευρά της μάχης. Θέλω να υπενθυμίσω ένα στοιχείο, ένα γεγονός σε όλους εδώ. Αν το Ηνωμένο Βασίλειο επιθυμεί ακόμα και τώρα να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τρόπο έφτακτο, αν αυτή είναι η επιθυμία του Ηνωμένου Βασιλείου, τότε αυτή η συνθήκη που διαπραγματευτήκαμε επί 1,5 χρόνο με την κυβέρνηση της Θερέζα Μέη, αυτή η συνθήκη είναι και θα παραμείνει η μόνη διαθέσιμη συνθήκη. Θα ήθελα αυτό να είναι ξεκάθαρο. Ακόμα μία φορά, δίπλα από αυτή τη συνθήκη, δουλέψαμε πάρα πολύ με την Βρετανική κυβέρνηση και κατ' εντολή και αίτημα τη βρετανική κυβέρνηση για να εξηγήσουμε, διευκρινίσουμε, εγγυηθούμε μέσω δύο εγγράφων επί των οποίων συμφωνήσαμε τη Δευτέρα το βράδυ. Εδώ, στο χώρο και στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Στρασβούργου. Η κυρία Μέη μας είπε ότι θα ήθελε να δηλωθεί, να δημοσιευθεί από πλευράς της μία μονομερής δήλωση. Τη Δευτέρα, σε αυτή την τελευταία συζήτηση που έγινε με την Βρετανική κυβέρνηση, θέλουμε να δώσουμε στην Βουλή των Κοινοτήτων, στο Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου, νέε διαβεβαιώσει, νέε διευκρινήσει για ένα συγκεκριμένο σημείο που είναι ο προσωρινό χαρακτήρα του μηχανισμού ασφαλεία του λεγόμενου backstop. Κάναμε το καταδύναμη. Ό,τι μπορούσαμε για να βοηθήσουμε την Βρετανική κυβέρνηση να πετύχει την στήριξη τη Βουλή των Κοινοτήτων με μόνιμο μέλημα, το οποίο εξέφρασα και εξ ονόματό σα. Να διαφυλάξουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ίσο τη Ιρλανδία. Να σεβαστούμε καθ' ολοκληρία την συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής και της συμφωνίας δηλαδή, του Belfast και να διασφαλίσουμε την ακαιρεότητα της εσωτερικής αγοράς μας, που είναι η αγορά όλων των 28 χωρών σήμερα και όσον ούπο των 27. Να διατηρήσουμε δηλαδή την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων υπέρ των καταναλωτών, δηλαδή διατροφική ασφάλεια, ασφάλεια των τροφίμων, οποιοδήποτε κίνδυνο να τον αποτρέψουμε για την ανθρώπινη υγεία. Ε, επίσης, υπάρχουν για τα, τους τελωνιακούς δασμούς, ε, για να υπάρχει ασφάλεια για τις επιχειρήσεις, ε, για να μπορούν να σέβονται ε, τους κανόνες και τα πρότυπα των εισαγόμενων προϊόντων. Η Βόρεια Ιρλανδία δεν είναι ένα θεωρητικό ερώτημα, δεν είναι ένα δόγμα δεν είναι το θέμα να δείξουμε ευελιξία. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ άμεσο και πρακτικό που αφορά την Ιρλανδία και την ειρήνη στην Ιρλανδία, η οποία θα πρέπει να είναι οριστική και που αφορά την προστασία τη εσωτερική αγορά. Οποιαδήποτε, οποιοδήποτε εμπόρευμα, οποιοδήποτε ζωντανό ζώο που μπαίνει από την Βόρεια Ιρλανδία μετά τον Brexit και που προέρχεται ε, ε από, την, ε, από το Ηνωμένο Βασίλειο, μπαίνει μετά στη Σλοβενία, στην Πολωνία, ε, στην Γερμανία, σε οποιαδήποτε από τις χώρες μας. Μια και έχουμε μια αγορά και, μια, και δεν υπάρχουν σύνορα. Θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο και θα προσπαθήσουμε να το καταφέρουμε να καταστήσουμε λειτουργικούς αυτούς τους ε, ελέγχους για τους καταναλωτές, για τον προϋπολογισμό και για τις επιχειρήσεις, έτσι, χωρίς να δημιουργήσουμε σκληρά σύνορα. Για τη χθεσινή ψηφοφορία διαπίστωσα ότι κάποιοι βουλευτές θέλουν ένα δεύτερο δημοψήφισμα, άλλοι προτιμούν το no deal, τη μη συμφωνία. Θεωρούν ότι αυτές οι νέες ε, νομικές εγγύησεις δεν αρκούν που βρήκαμε στη συζήτηση με την Τερέζα Μέη. Αυτές οι εξηγήσει και αυτές οι εγγυήσει ήταν σημαντικές. Και τη συμφωνήσαμε Δευτέρα βράδυ με τη στήριξη της Βρετανικής κυβέρνησης. Ο πρόεδρος Γιούνκερ το είπε πάρα αυτά, ότι δεν θα υπάρχει ερμηνεία ή εγγύηση περαιτέρω αυτών. Δεν μπορούμε να πάμε πιο πέρα. Συμπερασματικά θα να πω δύο λόγια για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Πού φτάσαμε σήμερα, πού είμαστε σήμερα το πρωί η ψηφοφορία που έχει αναγγελθεί από την Πρωθυπουργό για το, τη μη συμφωνία, το no deal. Σήμερα το βράδυ θα γίνει η ψηφοφορία αυτή και για την πιθανότητα παράταση που θα ψηφοφορήσει που θα λάβουν χώρα στη Βουλή των Κοινοτήτων. Μετά τι προφορίε αυτέ, η Βρετανική κυβέρνηση θα μα πει και ελπίζουμε θα μα το πει θετικά πώς επιθυμεί να προχωρήσει ούτω ώστε να υπάρξει μια επικοδομητική πλειοψηφία επί μιας πρότασης. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αυτή την ευθύνη πρέπει να μας πει τι θέλει για τη μελλοντική μας σχέση. Τι επιλογή κάνει. Όπως είπε και ο υπουργό, ποια είναι η ξεκάθαρη γραμμή που θα ακολουθηθεί. Αυτό είναι το ερώτημα που μπαίνει τώρα και που περιμένουμε μια απάντηση σε αυτό. Πάνω σε αυτό το ερώτημα που τίθεται, πριν από την απόφαση για πιθανή παράταση. Το να παρατείνουμε αυτή τη διαπραγμάτευση, να το κάνουμε. Αλλά γιατί μια και η διαπραγμάτευση για το άρθρο 50 έχει ολοκληρωθεί. Έχουμε τη συνθήκη. Είναι έτοιμη. Είναι εδώ. Περιμένουμε λοιπόν, αν τεθεί αυτό το ερώτημα, την απάντηση. Θα ήθελα να τα πω όλα αυτά και τα λέω σε μια πολύ σοβαρή χρονική στιγμή, γιατί ο κίνδυνος ε, της αποχώρησης χωρίς συμφωνία ποτέ δεν ήταν τόσο υψηλός. Μπορεί να βγει κατά τύχη και χωρίς συμφωνία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με άτακτο τρόπο το Ηνωμένο Βασίλειο. Να μην υποτιμήσετε παρακαλώ αυτό τον κίνδυνο, ούτε τις συνέπειές του. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι τους καλούμε με κάθε σοβαρότητα να προετοιμαστούν και από πλευράς της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και ο πρόεδρος Γιούνκερ έχει δώσει σαφείς οδηγίες και όλα τα κρατημέλη, χάρη στη δουλειά που κάνουν όλες οι προεδρίες και η δικιά σας κυρία Υπουργέ, ετοιμάζονται γι' αυτό. Δεν θέλουμε αυτό το σενάριο. Ποτέ δεν θέλαμε για να πριτανεύσει αυτή η επιλογή. Να αποχωρήσει χωρίς συμφωνία δηλαδή. Ναι, επικρατήσει το no deal. Όχι, θέλαμε πάντα μία έφτακτη αποχώρηση. Αλλά είμαστε έτοιμοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτό το ενδεχόμενο, αυτή την περίπτωση. Εάν δεν υπάρξει άλλη λύση που συμφωνηθεί, λόγω της λειτουργίας των συνθήκων, κατά ανάγκη θα βρεθούμε ενώπιον αυτού του νέου deal. Μερικές φορές, ακόμα και σήμερα το πρωί, με ρωτάνε αν είμαι απογοητευμένος, αν αισθάνομαι απογοήτευση μετά από αυτή την ψηφοφορία. Η απάντησή μου είναι πάντα ίδια. Σεβόμαστε το Ηνωμένο Βασίλειο και το λαό του είμαστε αποφασισμένοι, ήρεμοι και ενωμένοι και θα παραμείνουμε έτσι μέχρι το τέλος αυτής της εντυπωσιακή διαπραγμάτευσης. Θα υπερασπιστούμε τα συμφέροντα όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή θα είναι η γραμμή της διαπραγμάτευσής μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μισελ. Είσαι και διαπραγματεύτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, άρα σε ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και την ομάδα εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που την συντονίζει ο Γκί Φερχόφστατ και όλα τα μέλη της ομάδας αυτής για τη δουλειά που κάνουν για να επιλύσουν αυτό το τόσο σοβαρό και περίπλοκο πρόβλημα. Και τώρα περνάμε στις παρεμβάσεις των πολιτικών ομάδων. Ο Μάνφρεντ Βέμπερ, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, έχει το λόγο. Πρόεδρε, κυρία την Πρόεδρε, Μισελ, ε, κύριε εκπρόσωπε του Συμβουλίου, τι καταστροφή η χθεσινή ψηφοφορία. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω μια εντύπωση που είχα στο πόρτο της Πορτογαλίας. Συνομίλησα με νέους ανθρώπους οι οποίοι είχαν εργαστεί για λίγα χρόνια στο Λονδίνο. Έφυγαν ε, από την Πορτογαλία μετά από τα, οικογενειακά, τα οικονομικά προβλήματα. Συγγνώμη. Ε, επέστρεψαν όμως στην Πορτογαλία λόγω της αβεβαιότητας ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο και μας μίλησαν για τους φίλους τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μας είπαν πόσο δυσαρεστημένοι απελπισμένη είναι η ε, νεολαία στη Βρετανία, πόσο απογοητευμένη από την πολιτική του τάξη. Μια ολόκληρη γενιά θα υποφέρει, θα έχει λιγότερες ευκαιρίες για το μέλλον. Μια ολόκληρη γενιά δεν θα έχει τα ίδια ωφέλη με τις προηγούμενες γενιές. Μια ολόκληρη γενιά θα είναι θύμα της πολιτικής τάξης στο Λονδίνο. Γι' αυτό το πρώτο μου μήνυμα είναι ότι εμείς το, οι Ευρωπαίοι είμαστε στο πλευρό των νέων του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν θα σας αφήσουμε μόνους. Αυτό είναι το πρώτο μου μήνυμα. Το δεύτερο είναι τι κάνουμε τώρα. Σίγουρα πρέπει να προετοιμαστούμε για το χειρότερο σενάριο. Δεν μπορούμε να σώσουμε τους Βρετανούς. Εκείνοι πρέπει να αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν. Πρέπει να προετοιμαστούμε για το χειρότερο ενδεχόμενο. Το άλλο είναι ότι όταν αποτύχει η πολιτική τάξη, το λογικό επόμενο βήμα είναι να ξαναρωτήσει κανείς τους πολίτες. Και η τρίτη επιλογή είναι παράταση. Παράταση όμως με τι στόχο. Χρειαζόμαστε σωστά επιχειρήματα για να δώσουμε οποιαδήποτε ε, παράταση. Και γι' αυτό ας είμαι σαφής από πλευράς του ΕΛΚ. Δεν υπάρχει ανάγκη ούτε για μία μέρα παράτασης εάν δεν ξεκαθαρίσει η Βρετανική πλευρά τι θέλει να πετύχει. Αυτές λοιπόν είναι οι τρεις επιλογές που έχουμε. Θα ήθελα να προσθέσω ένα τρίτο σημαντικό στοιχείο. Ένα τείχος πυροπροστασίας. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ σαφή θέση χάρη στις εργασίες ε, των διαπραγματευτών της. Ε, είμαστε ενωμένοι, γνωρίζουμε τι ακριβώς θέλουμε, είμαστε σαφείς. Υπάρχει όμως ο κίνδυνο μέσα στις επόμενες εβδομάδες η πολιτική αβεβαιότητα στο Λονδίνο να επηρεάσει και την ευρωπαϊκή διαδικασία λήψη αποφάσεων ε, και έχω δύο πτυχέ κατά νου. Ε, από τη μία ξανασυζητάμε στο ε, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Brexit και όχι την Κίνα, τον ε, Τραμπ, ε, το διεθνές εμπόριο, όχι τα θέματα που είναι σημαντικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε να γεμίσουμε το πολιτικό χώρο μόνο με ε, το θέμα του Brexit λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας στο Λονδίνο. Και επίσης επίκυνται οι ευρωπαϊκές εκλογές. Ήδη κάποιοι από εμά έχουμε ξεκινήσει την προεκλογική εκστρατεία. Πρέπει λοιπόν να δείξουμε ότι αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι θα αποφασίσουν για το μέλλον τους. Δεν μπορούμε λοιπόν ε, να ε, ε, να γεμίζει ο πολιτικό χώρο από την πολιτική αβεβαιότητα στο Λονδίνο. Ελπίζουμε λοιπόν στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ξεκαθαρίσουν τι θέλουν. Για ε, πολλούς ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, οι εξελίξεις αυτές αποτελούν συναγερμό. Βλέπουμε τις πολιτικές εξελίξεις στο Λονδίνο και Όσοι δεν θέλουν να ακολουθήσουν τα βήματα αυτά θα πρέπει να καταπολεμήσουν το λαϊκισμό και την ε, παραπληροφόρηση. Ε, το Brexit είναι ε, προϊόν ακριβώς της παραπληροφόρησης και του λαϊκισμού. Θα πρέπει λοιπόν στην Ευρώπη να δημιουργήσουμε μια ισχυρή εταιρική σχέση για το μέλλον αυτής της Υπήρου, διότι πιστεύουμε στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Σας ευχαριστώ πολύ τώρα ο πρόεδρος των σοσιαλιστών, Ούντο Μπούλμαν, έχει το λόγο. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το Ανοιξιώτικο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνήθως είναι το η ευκαιρία να συμφωνήσουμε σχετικά με την οικονομική κατάσταση της Ένωσης. Σήμερα το πρωί μιλήσαμε για την αλλαγή του κλίματος. Έχω μία έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προς ε, την εκπρόσωπο του Συμβουλίου. Δεν απομένει χρόνος το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να γίνει Συμβούλιο Βιωσιμότητα. Ο Χάν Τίμερμαν έχει δίκιο. Δεν επιτρέπεται να περιμένουμε όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος. Πρέπει να εξετάσουμε τι εργαλεία έχουμε στη διάθεσή μας. Θα πρέπει το Σύμφωνο σταθερότητα και Ανάπτυξης να γίνει Σύμφωνο Βιωσιμότητα. Ε, θα πρέπει Ε, τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας να γίνουν μέσα βιωσιμότητα. Αυτό θα πρέπει να είναι το μήνυμα ε, τούτη την Άνοιξη. Και θα παρακαλούσα όσους έχουν επιρροή να την ε, εκμεταλλευτούν ώστε να έχουμε αυτήν την αλλαγή προτύπου που χρειαζόμαστε. Ο Αντώνιο Γκουτέρες ε, πριν 20 ε, χρόνια ξεκίνησε μια διαδικασία. Σήμερα είναι Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Ε, η οικονομία, οικολογία, κοινωνική συνοχή, ανταγωνιστικότητα τα συνδύασε. Δύο δεκαετίες έχουμε χάσει. Πρέπει όμως επιτέλους να αρχίσουμε να τα σκεφτόμαστε αυτά όλα μαζί. Και Βέιμπερ Εάν νέοι από το Λονδίνο επιστρέφουν στην Πορτογαλία, τότε αυτό έχει να κάνει με την ε, ανάπτυξη στη χώρα αυτή. Ο Αντώνιο Κώστα, ε, επικεφαλής της κυβέρνησης στην Πορτογαλία, με πολιτική κοινωνικής συνοχής και ε, οικονομικού εξυγχρονισμού και περιβαλλοντικής πολιτικής έχει καταφέρει να αποκαταστήσει την καλή κατάσταση της οικονομίας τέτοια, τέτοιου είδους μετασχηματισμό χρειαζόμαστε. Οι κοινωνίες μας χρειάζονται νέα ενέργεια, χρειάζονται ε, οξυγόνο, χρειαζόμαστε νέες ιδέες, να είμαστε προετοιμασμένοι για τέτοια. Δεν, θα χρειάζεται καν να ασχολούμαστε με το Brexit. Αυτή είναι η απάντηση στο Brexit, άσχετα από το τι θα γίνει συγκεκριμένα όσον αφορά τις τεχνικές λεπτομέρειες. Αυτή θα πρέπει να είναι η ευρωπαϊκή απάντηση στο Brexit. Νέα τόλμη, μια νέα ιδέα υπέρ των πολιτών και όχι εναντίον τους. Αυτό, αυτή είναι η καρδιά του προγράμματος που στηρίζουμε εμείς οι σοσιαλδημοκράτες. Μπορούμε όσον αφορά το Brexit μόνο να κάνουμε την έκκληση η Βουλή των ε, Κοινοτήτων ε, να αποτρέψει ένα σκληρό Brexit χωρίς συμφωνία από εκεί και πέρα όλα τα άλλα θα πρέπει να αποτελέσουν απόφαση των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου. Θέλουμε το, το Ηνωμένο Βασίλειο να παραμείνει κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν όμως κάτι τέτοιο δεν λειτουργήσει, εάν το Κοινοβούλιο παραμείνει μπλοκαρισμένο, τότε θα χρωστάμε κάτι στους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου ξαναπάρτε τον έλεγχο στα χέρια σας. Αυτό σημαίνει, η κυρία Μέη, ότι θα πρέπει οι πολίτες να έχουν την ευκαιρία να λάβουν νέα απόφαση, διότι το δικό τους μέλλον διακυβεύεται και όχι μόνο το μέλλον των βουλευτών. Αυτό θα πρέπει να τεθεί στο θεματολόγιο, αυτό θα πρέπει να συζητηθεί στην Σύνοδο Κορυφής. Θα πρέπει λοιπόν δύο σημαντικά θέματα να συζητηθούν. Ε, οι ευρωεκλογές να είναι ελεύθερες και δίκαιες και ναι, είναι ε, σωστά αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα, αλλά ε, τα προαιρετικά μέτρα των ε, επιχειρήσεων του διαδικτύου δεν αρκούν και επίσης πρέπει να ξανατεθεί στο θεματολόγιο το μεταναστευτικό. Δεν επιτρέπεται να αφήνουμε ανθρώπους να πνίγονται στη Μεσόγειο χωρίς να κάνουμε τίποτα. Σα παρακαλώ, λοιπόν, φροντίστε να ξανατεθεί το θέμα αυτό στο θεματολόγιο. Σα ευχαριστώ. Από το ECR, ο κύριο Έγκελ. Κύριε σου είπατε ότι δεν υπάρχει κάποια καλύτερη λύση. Κύριε Μπαρνιέ. Είπατε ότι δεν υπάρχει κάποια άλλη συνθήκη εκτό από αυτή που είναι διαθέσιμη. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτό ισχύει. Νομίζω ότι υπάρχουν και καλύτερε λύσει. Η καλύτερη λύση είναι να παραμείνει η Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επιτρέψτε μου να σας πω πώς θα το πετύχετε αυτό. Πρώτον, πρέπει να σταματήσουμε ε, να την πέφτουμε εντό αγωγικών στο Λονδίνο. Υπάρχουν εδώ άνθρωποι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που συνεχώ κατακρίνουν το Λονδίνο. Και ο κύριο Φάρατ και ο κύριο Βερχόφσταντ. δεν υπάρχει διαφορά ουσιαστικά σε ό,τι αφορά την κριτική που ασκούν στο Λονδίνο. Εκεί συμφωνούν. Δεύτερον, η Επιτροπή επιτέλου θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι έχει ευθύνη για τον Brexit. Η Βρετανία δεν ήταν πάντα υπέρ τη ε, επικουρικότητα, ε, τη αποκέντρωση, τη ανταγωνιστικότητα. Οι ε, Βρυξέλλε συνεχώ καταπατούν αυτέ τι αξίε. Είναι σαν μια χώρα να θέλει και να μπαίνει σε μια ομάδα ποδοσφαίρου και τελικά εσεί να παίζετε γκολφ ή κάτι διαφορετικό. Ποιο φταίει τελικά. Από επιχειρηματική πλευρά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το Brexit δεν είναι καταστροφικό μόνο για τη Μεγάλη Βρετανία, είναι καταστροφικό και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η Μεγάλη Βρετανία είναι σήμερα ο μεγαλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αποχώρηση της Βρετανίας ισοδυναμεί με μία ε, αποχώρηση υποθετική 19 μικρομεσαίων χωρών. Α αναγνωρίσουμε επίση ότι η Μεγάλη Βρετανία στο Κοινοβούλιο πάντα ήταν υπέρμαχο και προασπιστή ε, τη ελευθερία, ε, τη ανταγωνιστικότητα και χωρί την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο μάλλον, ε, θα, δεν θα είναι ανταγωνιστική η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με άλλες περιοχές όπως η Βόρειος Αμερική, η Ασία, η Κίνα, η Ιαπωνία και ούτε καθεξής. Θεωρώ λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τώρα μια ιστορική ευκαιρία να κάνει κάτι, να βοηθήσει ε, τους Βρετανούς που είναι υπέρ της παραμονής ε, στο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διεξαγάγουν ένα δεύτερο δημοψήφισμα. Και οι Brexiteers, οι υπέρμαχοι της αποχώρησης, να αλλάξουν γνώμη. Και έτσι να, καταφε... να τους βοηθήσουμε να αλλάξουν γνώμη και να ε, μην ντροπιαστούν κιόλας. Πρέπει λοιπόν όχι μόνο να τους ε, υποστηρίξουμε, αλλά και να τους ε, παράσχουμε τη δυνατότητα παράτεσης, άνευ όρων. Δεύτερον, κάποια αυτονομία σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της μετανάστευσής τους. Και αυτό είναι το κόλπο που θα μεταπίσει τη Μεγάλη Βρετανία και θα καταφέρουμε έτσι να διεξαχθεί δεύτερο δημοψήφισμα για να παραμείνει η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η Ένωση ποτέ δεν θα είναι πλήρη χωρί τη Μεγάλη Βρετανία. Εξ ονόματο των Φιλελευθέρων, ο κύριο Βερχόφστατ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να πω στον κύριο Χένκελ ότι προσωπικά πάντα έλεγα ότι η αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν μια τόσο μεγάλη χώρα φεύγει από την Ένωση είναι πολύ δύσκολο να πούμε «Μα τι ωραία». Αντιθέτως, η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εγώ είμαι αρκετά βέβαιο ότι η επόμενη γενιά σε ορισμένε δεκαετίε θα αποφασίσει την επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη υπάρχει αυτή η νέα γενιά και αυτοί θα πάρουν μια διαφορετική απόφαση από την απόφαση που ελήφθη από αυτή την κυβέρνηση και από την πλειοψηφία σήμερα. Αλλά κύριε Χένκελ, σας καλώ να τα πείτε αυτά στους φίλους σας, στη δική σας πολιτική ομάδα, στο ECR, που αυτή είναι η μεγαλύτερη υπέρμαχη του Brexit εύκολα ε, επικρίνετε εμάς εδώ και εμένα προσωπικά και λέτε ότι δεν είμαστε υπέρ του Βασιλείου, το, που το αντίθετο ισχύει, αλλά από την άλλη δεν είστε ε, σε θέση να πείσετε τους ε, συναδέλφους σας και δεν είναι εδώ για να σας χειροκροτήσουν, από ό,τι βλέπω κανείς δεν είναι εδώ. Δεύτερον, η πραγματικότητα, κύριε Χιάνκελ, είναι η εξή. Όσοι ξεκίνησαν όλη την υπόθεση του Brexit, που ουσιαστικά ήταν μια προσπάθεια του Συντηρητικού Κόμματο, με το οποίο συνεργάζεται και όλοι και το γνωρίζετε και πολύ καλά, ήταν ουσιαστικά μια προσπάθεια ε, να ξαναπάρουν τον έλεγχο. Αυτό τον μεγάλο σλόγγαν ε, ε, τη εξαρτία αποχώρηση θεωρώ ότι πλέον η κατάσταση εκτροχιάζεται στο Ενωνο Βασίλειο. Όχι, δεν ξαναπαίρνω τον έλεγχο, τον χάνουν πλήρω πια. Και ο μόνος εύλογο τρόπος επίλυσης του ζητήματο, και δυστυχώ δεν αναφερθήκατε σε αυτό κύριε Χένκελ, είναι να υπάρξει διακομματική συνεργασία στο βρετανικό πολιτικό προσκήνιο. Όσο γίνεται πιο γρήγορα να υπάρξει μια συμβαστική λύση μεταξύ συντηρητικών και εργατικών. Πώς γίνεται να λυθεί ένα επαρξιακό πρόβλημα όπως το Brexit όταν και τα δύο κόμματα ε, αξιοποιούν ε, το Brexit ε, ο ένας κατά του άλλου. Για αυτούς είναι ένα όπλο στη φαρέτρα τους, όχι υπαρξιακό πρόβλημα. Επομένως, και η δική μας έκκληση αλλά και η δική σας στην Ολομέλεια δεν θα πρέπει να απευθύνεται σε εμά, αλλά προς το βρετανικό πολιτικό στερέωμα ότι πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία εξέβρεση συμφωνίας μεταξύ των δύο μεγάλων πολιτικών κομμάτων και να υπάρχει τελικά μία θέση την οποία να μπορούμε και εμείς να στηρίξουμε ή μία στενή συνεργασία μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι Ήτη διέξοδος. Και ουσιαστικά αυτό που χρειάζεται είναι η χώρα και η βασίλισσα να τεθούν ε, σε πρώτη θέση και να μην ε, εξυπηρετούν όλα τα συμφέροντα του ε, Βρετανικού Κοινοβουλίου. Φτάνω λοιπόν στο επόμενο ζήτημα. Παράταση. Εγώ δεν θέλω κάποια μακροπρόθεσμη παράταση. Σας το λέω ανοιχτά. Μια παράταση που θα υπερβαίνει τις ευρωεκλογέ, που τελικά οι ευρωεκλογέ δεν θα έχουν να κάνουν με τίποτα άλλο, με κανένα άλλο θέμα. Μόνο με το Brexit. Δεν θα μιλήσουμε για, για τα πραγματικά ζητήματα και τι πραγματικέ μεταρρυθμίσει που χρειαζόμαστε στην Ευρώπη. Και θα δώσουμε και ακόμα μία θητεία στον κύριο Φάρατζα, έτσι. Αυτό ακριβώ θέλει και εκείνο. Γιατί το θέλει, για δύο λόγου. Πρώτον, για να συνεχίσει να πληρώνεται, να έχει μισθό που θα μπορεί να μεταφέρει στην ε, offshore εταιρεία του. Και δεύτερον, Και δεύτερον, να συνεχίσει να κάνει τη βρωμοδουλειά του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, προσπαθεί να καταστρέψει την Ένωση εκ των έσω. Αυτό είναι ο πραγματικό του σκοπός. Δεν χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε σαφήνεια και βεβαιότητα από την Βουλή των Κοινοτήτων. Κάτι που ζήτησε ο κύριο Χένκελ. Αυτό χρειαζόμαστε. Είμαι κατά οποιασδήποτε παράταση, ακόμα και μία ημέρα ή μία εβδομάδα, 24 ωρών ακόμα. Είμαι κατά εάν δεν βασίζεται σε μια σαφή θέση της Βουλής των Κοινοτήτων. Να γνωρίζουμε ακριβώς τι θέλουν. Αν, ακόμα και αν είναι κάτι λιγότερο φιλόδοξο από την συμφωνία. Ακόμα και αν είναι συμφωνία για τελωνιακή ένωση ένα μοντέλο Νορβηγία Plus. Ό,τι θέλετε, αλλά πάρτε μια απόφαση στο Λονδίνο. Αυτή η αβεβαιότητα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ούτε για εμά ούτε για τη Βρετανία και σίγουρα όχι για του πολίτε μα. Ευχαριστώ. Τώρα το λόγο έχει ο πρόεδρο τη ομάδα των Πρασίνων, Φιλίπ Λαμπέρ. Ευχαριστώ πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ακόμα μια φορά. Ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αποφάσισε να σνομπάρει την Ολομέλεια. Είναι εντυπωσιακό στο βαθμό που οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων γενικά δεν τα έχουν πάει καλά. Πάντα συζητάμε άσυλο, μετανάστευση. Υποτίθεται ότι ο Ντόναλτ Τάσκ έχει προτεραιότητα αυτό το θέμα. Μετά από τρία χρόνια θα περιμέναμε λογικά κάπου το Συμβούλιο να αποφασίσει για αυτό το πρόβλημα. Το Συμβούλιο αποφάσισε όμως ότι δεν θα συμφωνήσει τίποτα μόλις τώρα. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων δείχνουν την αδυναμία τους ή την έλλειψη θέλησής τους να συνοηθούν. Χρειάστηκε ε, στο Κοινοβούλιο ε, να βρούμε μία πλειοψηφία δύο, τριών, ε, δύο τρίτων για την κοινή θέση. Εμείς τα καταφέραμε. Περιμένουμε ακόμα τους leaders, τους ηγέτες. Πού είναι όταν ο επιστημονικός κόσμος ματίνει μόνο 12 χρόνια, όχι περισσότερο, για να σώσουμε τον πλανήτη και το κλίμα. Για να σώσουμε τη βιοπικιλότητα. Ακόμα και εδώ οι leaders είναι τυφλοί, κουφοί και μουγγοί απέναντι στην οργή της Ευρωπαϊκής Νεολαίας. Περιμένουμε το Συμβούλιο να βάλει αυτό το, θέμα στην καρδιά των συζητήσεων. Όταν οι πολίτες ξεσηκώνονται για να αρνηθούν μια κοινωνία όπου ο πλούτος συγκεντρώνεται σε όλο και λιγότερα χέρια, πού είναι αυτή η αρχική, ε, όπου έχουμε ανισότητες λόγω των του φορολογικού ανταγωνισμού των κρατών μελών. Ε, λόγω του ότι ε, υπάρχει άγρια παγκοσμιοποίηση. Θέλουμε οι leaders να το συζητήσουν αυτό το θέμα. Αλλά δεν έχουν, το έχουν συνειδητοποιήσει καν. Πού είναι η ηγετική δύναμή τους και ρόλος τους. Όλο και περισσότεροι leaders επιλέγουν να υποσκάψουν τα θεμέλια της δημοκρατίας μας. Το διαχωρισμό των εξουσιών ανεξαρτησία της ε, δικαιοσύνης, του τύπου, σεβασμός της ε, ιδιωτικότητας, της ε, αναλογικότητας ή την κατάπνιξη της βίας, την κατάπνιξη μάλλον των διαδηλώσεων με τη βία. Τον Ιούνιο στο Συμβούλιο υποτίθεται θα πρέπει να ξεκινήσει μία διαδικασία κατά της Ουγγαρίας. Περιμένουμε, κυρία μου, κάτι παραπάνω από μία ευγενική απάντηση. Επίσης, το Brexit θα πρέπει να σταματήσουμε να μας διασκεδάζει ε, και να απλώς έτσι να ξεχνούμε τα βασικά θέματα. Περιμένουμε τους leaders να γίνουν leaders και όχι ακόλουθοι. Η πραγματική ηγεσία είναι να διατηρήσουμε το περιβάλλον, να υπάρξει κοινωνική δικαιοσύνη, να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και τις ελευθερίες μας και να το βάλουμε στην ε, καρδιά της πολιτικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωση και της φιλοδοξία. Τη. Ευχαριστώ. Και τώρα, η πρόεδρος της ομάδας της ΓΚΟΕ, η κυρία Τσίμερ, έχει το λόγο. Κυρίες και κύριοι, ε, νομίζω ότι όλοι γνωρίζετε την ταινία «Η μέρα της Μαρμότας». Αυτό ζω κι εγώ κάθε φορά που σκέφτομαι το επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου πάλι θα δεσπόσει η συζήτηση για τις συνέπειες του Brexit και τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχουν εδώ όμως σημαντικά θέματα η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοστάτησε στην επίτευξη της Συμφωνίας του Παρισιού. Πρωτοστάτησε ε, όσον αφορά την ε, συνθήκη βιωσιμότητας. Αλλά αυτά είναι τα θέματα που θα πρέπει να μας απασχολήσουν, διότι έτσι θα μπορέσουμε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να πετύχουμε στόχους, λαμβάνοντας υπόψη και τα όσα συμβαίνουν εκτός των συνόρων μας. Ε, έτσι θα εξασφαλίσουμε αξιοπρεπή διαβίωση για τους πολίτες μας, αλλά και για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Αυτό θα πρέπει να πετύχουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανταυτού όμως ε, για δεύτερη φορά είδαμε αποτυχία της συμφωνίας στην Βουλή των Κοινοτήτων σε, σε τείχο προσέκρουσε η Τερίζα Μέη. Δεν ε, έχουμε πλειοψηφία για μια συντεταγμένη αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η κατάσταση. Τις ε, συνέπειες ε, θα τις υποστούν ε, καταρχάς ε, οι πολίτες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και οι Ιρλανδοί. Πολύ... πολλές επιχειρήσεις θέλουν να μεταφέρουν ε, την ε, έδρα τους ε, στο Belfast θεωρώντας ότι η Ιρλανδία θα παραμείνει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πολλοί δεν έχουν τη δυνατότητα να μετικήσουν. Πολλοί έχουν ζητήσει ε, υπηκότητα άλλου κράτους μέλους. Ε, οι περισσότεροι όμως δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή και θα νιώσουν τις συνέπειες στην πρόσβασή τους στα συστήματα υγείας, ε, στην εκπαίδευση, στις οικονομικές και διαρθρωτικές συνέπειες για τις περιοχές τους. Και αυτού θα πρέπει να σκεφτούμε, τους πολίτες, όχι την κυβέρνηση ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, όχι την Βούλη των Κοινοτήτων. Αυτή είναι η υποχρέωσή μας. Τους πολίτες πρέπει να σκεφτούμε. Και δύο συνέπειες θα πρέπει να συζητήσουμε. Θα πρέπει να συζητήσουμε τις ε, συνέπειες ε, μιας ε, αποχώρησης στις 29 Μαρτίου. Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των πολιτών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι η υποχρέωσή μας. Έχουμε αναλάβει μια ευθύνη και θα πρέπει να το δηλώσουμε αυτό με σαφήνεια. Και θα πρέπει επίσης να υποστηρίξουμε σαφώς την Ιρλανδία και να πούμε ότι είμαστε κατά σκληρού συνόρου και κατά οποιασδήποτε τροποποίησης της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής. Δεν επιτρέπεται να διακυβευτούν τα δικαιώματα των πολιτών ε, σε αυτά τα μέρη της Ευρώπης. Υπάρχει όμως μία λύση ε, για το θέμα του backstop. Να μην υπάρχουν ε, σύνορα στο νησί της Ιρλανδίας. Η Ιρλανδική ενοποίηση θα ήταν η πιο απλή λύση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είχε πρόβλημα. Ε, η Ιρλανδία δεν θα είχαν πια πρόβλημα. Και όσοι επιθυμούν το Brexit σίγουρα δεν θα είχαν πρόβλημα. Μήπως ε, μία μικρή ε, Μεγάλη Βρετανία είναι πιο σημαντική για την ε, Τερίσα Μέη ε, από την παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δούμε αν εννοεί στα σοβαρά τα λόγια της. Ευχαριστώ πολύ. Από το EFDD ο Νάιτζελ Φάρατζ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μετά από σχεδόν 20 χρόνια, πραγματικά ελπίζω να είναι η πρώτη τελευταία μου ομιλία σε αυτό το κοινοβούλιο και να μην ξανάρθω εδώ τον Ιούλιο. Και είμαι σίγουρος ότι πολλοί θα συμφωνήσετε μαζί μου. Σα είπα, κυρία Μπαρνιέ, ότι αυτή η συνθήκη δεν θα περνούσε από το Κοινοβούλιο. Δεν με πιστέψατε, καταψηφίστηκε. Νομίζω ότι το παρατραβήξατε, ζητήσατε πάρα πολλά. Και σήμερα το πρωί βρίσκεστε ε, φτωχότερους κατά 39 δις ε, λίρες. Δεν ξέρω αν σας αρέσει αυτό, αλλά μην ανησυχείτε. Θα σας βοηθήσουμε, γιατί σήμερα το Κοινοβούλιο θα κάνει ό,τι μπορεί για να προδώσει την ε, ψήφο υπέρ της αποχώρησης. Το άρθρο 50 λέει ότι πρέπει να φύγουμε στις 29 Μαρτίου με ή χωρίς συμφωνία. Και πρέπει να σα πω ότι αυτή τη στιγμή το κενό, το χάσμα μεταξύ του πολιτικού στερεώματο στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη κοινή γνώμη είναι χαόδη. Γιατί η κοινή γνώμη είναι ενωμένη εδώ και χρόνια στη χώρα μου. Θέλουμε να φύγουμε. Είναι πολύ απλό. Και αυτό ισχύει και για πολλούς που ψήφισαν υπέρ της παραμονής, γιατί ακριβώς υπερασπίζονται την αρχή της δημοκρατίας. Ως εδώ Έχουμε δει ε, ε, όλη αυτή την ε, κακιασμένη και θυμωμένη αντίδραση του κυρίου Βερχόφστατ απέναντί μου, του κυρίου, απέναντί μας μάλλον, του κυρίου Μπαρνιέ, του κυρίου Τίμερμαν, του κυρίου Τούσκ. Και δεν θέλουμε να συνεχίσετε να μας κυβερνάτε. Θέλουμε εμείς να ορίζουμε τη μοίρα μας. Είμαι σίγουρος ότι στα επόμενα επεισόδια η κυρία Μέη θα, θα πάει στις Βρυξέλλες